Good morning. Καλημέρα σας. Φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε. Παρακαλώ καθίστε. Πρώτο θέμα τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών χθες το βράδυ. Πληροφορήθηκαν οι συντονιστές για το πρόγραμμα της πρώτης δημόσιας ακρόασης περί της πρωτοβουλίας των πολιτών που θα οργανωθεί 17 Φεβρουαρίου Δευτέρα στις 3. Εδώ και αρκετό καιρό είχαμε στείλει ένα έντυπο στους ενδιαφερόμενους για να εγγραφούν και είχαμε διανύμει και το πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα σε συμφωνία με την Επιτροπή Περίφ που είναι και η αρμόδια για αυτή την ακρόαση. Πήραμε μερικές απαντήσεις και όλοι όσοι ενεγράφησαν θα συμμετάσχουν καταλήλως. Δεύτερον, το, ιστόθυρα web της Επιτροπής μας. Από το 2010 προσπαθήσαμε να οργανώσουμε αυτό το επικοινωνιακό εργαλείο που θα βοηθήσει ελπίζουμε την επαφές, επαφές μας με τους πολίτες. συνεννοηθήκαμε και με ομάδες και υπηρεσίες για να είναι όλα έτοιμα μέχρι το τέλος της θητείας ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στους διαδόχους μας στην Επιτροπή εδώ το εργαλείο αυτό έτοιμο. Επίσης και άλλες δραστηριότητες προβλέπονται τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε στις προτάσεις που έχουμε λάβει. Τις επόμενες μέρες και ελπίζουμε πριν τελειώσει η θητεία να έχουν καταλήξει όλα αυτά. Τώρα για το σημείο 3 οι συντονιστές Γιάρ και Μποστινάρου μας θύμισαν ότι έχουν την πρόθεση να αποστείλουν επιστολή στο Γενικό Γραμματέα κύριο Βέλε για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας της Επιτροπής μας. Οι συντονιστές το έλαβαν υπόψη, το σημείωσαν δηλαδή, αν και μερικοί διαφωνούσαν με την ίδια την επιστολή και επομένως η πρωτοβουλία αυτή παραμένει πρωτοβουλία των δύο που την πρότειναν. Τώρα, για τις δύο επόμενες συνεδριάσεις μας πριν λήξει η θητεία, θα συμπληρώσουμε την ημερήσια διάταξη ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τις ημερήσιες αυτές διατάξεις από πριν σε συνεννόηση με τους συντονιστές. Τη αιτήση των Μποστινάρου, Πάσκα και Σαλαβράκου οι συντονιστές αποφάσισαν με πλειοψηφία να αλλάξουν τη σύσταση για την αναφορά 1002-2013 που θεωρείται τώρα πλέον απαράδεκτη. Όσο για το αίτημα του συναδέλφου Ινάγκη να τροποποιηθεί η σύσταση για την αναφορά 866-13 και να θεωρηθεί αποδεκτή, με την ίδια πλειοψηφία οι συντονιστές δέχτηκαν την πρόταση αυτή του συναδέλφου μας Φερνάντε Σινάκη. Στο 3 τώρα, ε, στο 6 για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή περί Frontex. Σας υπέβαλα, σας έστειλα το αίτημα της διάσκεψης των Προέδρων, αλλά δεν κατέληξε. Και η άσκεψη δηλαδή δεν δέχτηκε αυτή την ειδική έκθεση που είχαμε ζητήσει και, είχε ζητήσει, και πράγμα το οποίο είχε ζητήσει και ο διαμεσολαβητής. Η συνάντηση των συντονιστών αποφάσισε επίσης να γραφτεί ειδική έκθεση από την Επιτροπή μας και θα αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσει να συνταχθεί αυτή η έκθεση. Τώρα για τα αιτήματα κατεπίγοντος, ε, δηλαδή άδειες που είχαν ζητηθεί από την περασμένη συνεδρίαση, διανύμαμε έναν κατάλογο αιτημάτων κατεπίγοντος που εξέτασαν και οι συντονιστές με τη γραπτή διαδικασία. Εχθές ζητήθηκε αναθεώρηση ορισμένων γνωμοδοτήσεων για τέσσερα νέα κατεπήγοντα που μας είχαν ζητηθεί από τους πράσινους. Για τα αιτήματα αυτά είπαμε ότι θα αποφασίζαμε εν καιρό το δέοντι με γραπτή διαδικασία, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή. Επίσης μοιράστηκε ένα γράμμα, επιστολή και παρακαλώ να τη διαβάσουν εδώ όλα τα μέλη, είναι επιστολή του Επιτρόπου Μπαρνιέ για την επικύρωση της συνθήκης του Μαρακές που αφορά άτομα με αναπηρίες και ξέρετε ότι παίζουμε σημαντικό ρόλο και εμείς. Είμαστε από τους κύριους συνομιλητές από αυτού του Μπαρνιέ και της Επιτροπής γενικότερα. Έχει διανεμηθεί, διαβάστε το και αυτό, γιατί συνοψίζει και ενημερώνει τις δραστηριότητές μας με όλες τις αναφορές που έχουν ληφθεί, εκείνες που εξετάζονται και εκείνες που ακόμη πρέπει να εξεταστούν. Για να γνωρίζετε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Δεν έχει αποφασιστεί τίποτε άλλο. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, τότε το αποτέλεσμα της συνεδρίας των συντονιστών εγκρίνεται. Δεν έχει ζητηθεί κανένα λόγος από κανέναν, άρα εγκρίνεται μια στιγμή, μια στιγμή να ελέγξω εδώ κάτι που μου λένε Περνάμε στο επόμενο σημείο δηλαδή στην ψηφοφορία. Έχουμε τρία έγγραφα προς ψήφιση. Το πρώτο είναι η έκθεση 2013 για την Ιθαγένεια της Ένωσης. Η συγητής είναι ο κύριος Σαλαβράκος. Και του δίνω αμέσως το λόγο πριν την ψηφοφορία αν θέλει. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και και όλους τους συναδέλφους διότι νομίζω ότι καταλήψαμε σε ένα κείμενο το οποίο είναι αρκούντος αποδεκτό από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαβράκο. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία για το ψήφισμα 2013 για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ενωσιακή Ιθαγένεια του κυρίου Σαλαβράκου. Ο Μποστινάρου προτείνει να δούμε αν λειτουργούν εμιχανέ. Να επαναβαληθεύσουμε λοιπόν. Δοκιμαστική ψηφοφορία λοιπόν 16 18 ψήφισαν συνολικά. 16 υπέρ 2 κατά βγήκε. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πιο πολλοί από 18. Ποιος δεν ψήφισε. Α, εσείς. Α, μάλιστα. Μάλιστα. και η κυρία Βέρτμαν, δηλαδή 20 είμαστε που ψηφίζουμε, εντάξει. Αρχίζουμε λοιπόν. Αρχίζουμε με τη συμβιβαστική 1. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρέπει όμως να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Δεύτερο τμήμα. Περ, κατά, αποχές. Απαρρίπτεται αλλά θα το επαληθεύσουμε. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 3. Όχι της τροποπολογίας 43, ε, γνώμη λέει η πρόεδρος. Έληξε. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά χές εγκαρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά χες εγκρίνεται τροπολογία 28 υπέρ κατά χες εγκρίνεται τροπολογία 30 υπέρ κατά χες απορρίπτεται Ανθρωπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά ψυχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 με προφορική τροποποίηση είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης όχι τότε μπορούμε να ψηφίσουμε την 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά εποχές επαλήθευση 73 απορρίπτεται ισοψηφία 9-9 με δύο αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απαρρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης. Όχι. Σε δύο τμήματα λοιπόν. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, να επαληθεύσουμε για το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα. Ήταν σαφές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εφτά υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 με προφορική τροποποίηση είναι κάνει κατά της προφορικής τροποποίησης ψηφίζουμε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έντεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 με προφορική τροποποίηση είναι κανείς κατά όχι 16 υπέρ κατά δεν είναι σαφές επαλήθευση ηλεκτρονικά για τη 16 15 με 6 εγκρίθηκε λοιπόν. 18 υπέρ. Κατά. Ποχέ απορρίπτεται. Ναι, 19 υπέρ. Κατά. Ποχέ. εγκρίνεται. 20 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά. Όχι. 20 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 21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 ηλεκτρονικά άρχεται έληξε ομόφωνη έγκριση μεγάλη επιτυχία του κυρίου Σαλαβράκου ευχαριστούμε και πάλι κύριε Σαλαβράκο για την εξαιρετική εργασία σας. έκθεση 2013 δραστηριότητων της Επιτροπής. Ο κύριος Βαλένσα δεν θέλει να λάβει το λόγο. Ας πάρω μια ανάσα και ας προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής των Αναφορών 2013. Τροπολογία 23. Πέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 4 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 23. Η 24 παρακαλώ υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά άποχες δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι για να σας βλέπω καθαρά αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία στην 26 πέρας 20 υπέρ μία ψήφος κατά αναμφίβολα ενεκρίθη μάλλον δεν λειτουργεί καλά, δεν κάνει καλά τη δουλειά του διευθυντή τη ορχήστρα. Γιατί βλέπω να μην σηκώνετε με τρόπο συντονισμένο τα χέρια σα. Παράγραφος 4α. Νέα. Συμβιβαστική τροπολογία προφορική. Όχι, ζητώ συγγνώμη, γυρνάω πίσω στην 27. Υπέρ, κατά, Άποχες. Απερίφθη. Και τώρα η συμβιβαστική. Η προφορική συμβαστική τροπολογία μετά την παράγραφο 4α, νέα παράγραφος, την ψηφίζουμε, εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Προφορική. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Όχι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Ε, βλέπω εδώ ένα λάθος. 29 σε τρία τμήματα έχει γίνει ο χωρισμός σε τρία τμήματα για την 29. Υπάρχει ένα λάθος στον, ε, στις γραμμές που έχουμε χαράξει στον κατάλογο, γιατί βλέπετε μια διαχωριστική γραμμή, αλλά πρόκειται για την ίδια τροπολογία, 29 σε τρία τμήματα. Ψηφίζουμε λοιπόν, το, ψηφίσαμε το πρώτο τμήμα, τώρα πάμε στο δεύτερο τμήμα. Της 29, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τρίτο τμήμα της 29, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Η 30 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 παρακαλώ, τροπολογία 40 υπέρ κατά Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε παρακαλώ την 40 ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. 10 υπέρ, 11 κατά, απερίφθη. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 43 43 Πέρας. Ομόφωνα. 21 υπέρ. 44 παρακαλώ. Ήταν τόσο σαφέ το αποτέλεσμα που δεν ήταν εμφανέ. 44 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχέ. Απερίφθη. 45 δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχέ. Απερίφθη. Όχι, εγκρίνεται, ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 19, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία, την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 οκτώ. Τρία τμήματα. Πρώτο παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 49 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη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 66 υπέρ κατά άποχες απεριφθεί 67 υπέρ κατά άποχες δεν είναι σαφές για μένα να το επαληθεύσουμε 67 παρακαλώ πέρασε Δεκάξι υπέρ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 αποχές απερίφθη. Τροπολογία 10. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές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 18 υπέρ, 3 κατά. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον κύριο Βαλέντζα. Now the last... Και τώρα η τελευταία ψηφοφορία όσον αφορά το έγγραφο εργασία για την ε, εξοπλιστική των πραγμάτων επιτροπή στην Ελλάδα. Ο κύριος Σιτουργκάη θα λάβει το λόγο, αν θέλει, πριν την ψηφορία, όχι. Οπότε τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία. Πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαρχμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπάρχει εδώ μια τεχνικού χαρακτήρα διόρθωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Με προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά όχι επομένως υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7. Με προφορική τροπολογία ενίσταται κανείς όχι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 με προφορική τροπολογία Κνήσατε κανείς, όχι, ψηφίζουμε την 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 με προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα. Είναι κανείς κατά της ε, προφορικής τροπολογίας, όχι. Επομένως, ας ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεύτερο τμήμα της 11, λέει η πρόεδρος. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσαμε το πρώτο. Μόλις το ψηφίσαμε το πρώτο. Και τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο. Η κυρία Παλιαδέλη λέει διότι απερίφθη το πρώτο. Οπότε τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο. Λέει πρόεδρος. Οπότε ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα του 11. Πέρα ψηφοφορίας 22 εγκρίνεται. Στο 13 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν σηκώνει κανείς όπως πρέπει το χέρι του για το 13. Πέρας. Για το 14 τώρα. Ε, απορρίπτεται. 15. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Με προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα. Προφορική τροπολογία και σε δύο τμήματα. Είναι κανεί κατά τη προφορική, όχι. Επομένω, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 17 με την προφορική τροπολογία. Είναι κανεί κατά. Μάλιστα, ο κ. εγώ έχω μία ένσταση. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω για αυτή την ε, ε, τροπολογία ότι ενίσταμε διότι ο λόγος πολιτισμού ομάδας θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλντίνη. Επομένως, θα ψηφίσουμε το 17 της ε, κυρία Σάουκεν όπως διατυπώθηκε. Ποιος είναι υπέρ, κατά, ποιος απέχει, εγκρίνεται το 18, είχε αποσυρθεί τροπολογία 19 με την προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας. Ουδής. Επομένως ψηφίζουμε το 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε. Chiudo la votazione. All'unanimità 22 voti a favore, complimenti al collega. Εγκρίνεται με 22 ε, ψήφους, ε, ψηφι ομοφωνία. Συγχαρητήρια κύριε Τουργκάη. Abbiamo così concluso. Οπότε τώρα ολοκληρώσαμε τι ψηφοφορίε. Έχουμε, όπως είπαμε χθες, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντο από την Ελλάδα. Οπότε τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Νιώκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νιώκας. Είμαι, εκπροσωπώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Είμαι συνεργάτης του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Μανιάτη και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την Επιτροπή και να αναφέρω ότι προσδοκούμε ότι με τις ε, ακριβοδίκες αποφάσεις της θα ενθαρρύνει τις μεγάλες προσπάθειες που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη στη χώρα μας όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και σημαντικό ακόμα δρόμο να διανύσει, ώστε να φτάσει στα απαιτούμενα επίπεδα, προκειμένου ως πολιτεία να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο κάθε πολίτης και κάθε παραγωγός αποβλήτων έχει πρόσβαση στο κατάλληλο σύστημα διαχείρισης. Έτσι κι αλλιώς αυτός έχει την ευθύνη των αποβλήτων του. Το Υπουργείο καταβάλει συστηματικές προσπάθειες αφενός να αντιμετωπίσει αδυναμίες και υποχρεώσεις από το παρελθόν και αφετέρου να προχωρήσει με συστηματικό σχεδιασμό και γοργά βήματα στην ουσιαστική αναβάθμιση του τομέα, στον αναπροσδιορισμό του και στην εφαρμογή των νεότερων κατευθύνσεων του κοινοτικού κεκτημένου. Είναι γνωστό ότι δεν τηρείται αυτή τη στιγμή η ιεράρχηση που προβλέπει η οδηγία στη χώρα μας, με δεδομένο ότι πάνω από το 80% σήμερα των αποβλήτων διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής και μάλιστα εξαλείφεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο εξαλείφεται η ανεξέλεκτη διάθεση η οποία ε, σε πολύ μικρό βαθμό απέμεινε. Ο λόγος που δεν τηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια η ιεράρχηση αυτή που σήμερα προσπαθούμε να την ανατρέψουμε είναι ότι ο μεγάλος αριθμός των ανεξέλεκτων χωματερών που είχαμε από το 2004 Ξέρετε ότι υπήρξε και καταδίκη της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2005 από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο μεγάλος αριθμός και η καταδίκη μας οδήγησε στην αντιμετώπιση, στην εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος δράσης για τη διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης και παράλληλα τη δημιουργία ενός δικτύου υποδομών υγειονομικής ταφής αυτή η τεράστια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε στο ότι οι 3.036 χωματερές που υπήρχαν το 2004 να έχουν αποκατασταθεί στη συντριπτική τους πλειοψηφία και σήμερα να έχουν απομείνει ελάχιστες γύρω στις 70 οι οποίες φυσικά είναι ενταγμένες όλες σε προγράμματα αυτή τη στιγμή αποκατάστασης γίνονται έργα και προσδοκούμε εντός του 2014 να έχουν αποκατασταθεί, αν όχι όλες, μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2015 θα έχουν ολοκληρωθεί. Όμως, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι η υγειονομική ταφή είναι στο τελευταίο σκαλί της ιεράρχησης και θέλουμε να το ανατρέψουμε, Ήδη στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, χθες μάλιστα στην Αθήνα υπήρξε μια μεγάλη εκδήλωση δημόσιου διαλόγου πάνω στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων σε εφαρμογή του πνεύματος και του γράμματος της οδηγίας ε, πλαίσιο για τα απόβλητα αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας του νόμου 4042 του 2012 και μέσα σε αυτό το σχέδιο τα πάντα αλλάζουν τα πάντα αλλάζουν εφαρμόζεται η ιεράρχηση που προβλέπει η οδηγία προτάσεται η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων η επαναχρησιμοποίηση η ανακύκλωση η ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας αφήνοντας στο τελευταίο σκαλί της ιεραρχίας τη διάθεση στους χιτά. Ήδη και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης ολοκληρώνεται και το, ε, τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων θα εναρμονιστούν με βάση τον εθνικό σχεδιασμό. Αναφέρω τρία χαρακτηριστικά ε, θέματα τα οποία δείχνουν ότι στην πράξη δεν είναι μόνο οι σχεδιασμοί που εφαρμόζονται αλλά στην πράξη τα πάντα αλλάζουν. Το ένα παράδειγμα είναι ότι έχουμε 15 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Έχουμε διαγωνισμούς σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων για τις 5 υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσωρινή ανάδοχοι και τα συμβόλαια προβλέπουν μέσα στους επόμενους 20 μήνες να κατασκευαστούν, ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της ανακύκλωσης στη χώρα μας, ότι έχουν γίνει, έχουν γίνει ενέργειες συμφωνίας εθελοντικής με βιομηχανίες όπως η τσιμεντοβιομηχανία για συναποτέφρωση και εφαρμογή της ενεργειακής αξιοποίησης ειδικά για το RDF για το οποίο μάλιστα επεξεργάζεται και αυτή τη βδομάδα υπογράφεται κοινή υπουργική απόφαση για τις προδιαγραφές χρησιμοποίησης απορριμματογενών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία και άλλες παρόμοιες βιομηχανίες. Με αφορμή και το EU Pilot που υπάρχει για την ανακύκλωση γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια έρευνας της ε, κατάστασης και της ε, βελτιστοποίησης της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Ε, ευχαριστώ. Είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε. Εμείς. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κίκα. Ένα λεπτό κύριε Κίκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτό, τι μπορώ να πει κανεί ένα λεπτό. Εγώ θα επικεντρωθώ στην προηγούμενη φορά όταν ήμουν παρόν εδώ ε, και άκουσα τα, τους κύριους ευρωβουλευτές. <clears throat> Α, μάλιστα τους είδα έτσι πολύ διστακτικούς και αναποφάσιστους ε, συζητήθηκε την προηγούμενη ε, συνεδρίαση στις 21 Ιανουαρίου η αρχή της επικουρικότητας. Ε, εγώ θα ήθελα να σταθώ ότι, και να πω ότι η αρχή της επικουρικότητας είναι η αρχή που ρυθμίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων. Πρέπει να επιτρέπει τον καθορισμό του κατά πόσο η Ένωση μπορεί να ενεργήσει ή πρέπει να αφήσει την πρωτοβολία στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η Ένωση μπορεί να παρεύει σε τομεί οι οποίε δεν επίπτουν την αποκλειστική τη αρμοδιότητα, παρά μόνο εάν και στο βαθμό που οι στόχοι τη προβλεπόμενη δράση και εδώ στην προκειμένη περίπτωση η διαχείριση είναι των απορριμμάτων, είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώ από τα κράτη-μέλη και δύναται συνεπώ λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων τη προβλεπόμενη δράση να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωση. Στην περίπτωση εδώ που μιλάμε υπάρχει το πρώτο σφάλμα. Θα πρέπει να Υπάρχει και η αρχή της πρόσληψης και, για αυτή, και βάσει αυτής της αρχής είμαστε εδώ και γι' αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Να, αποτρέψουμε το οικολογικό και οικονομικό σκάδο που συντελείται όχι μόνο για το γραμματικό αλλά για όλους τους χιτάς στην Ελλάδα. Είναι λίγο ο χρόνο, δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα. Ε, θα επικεντρωθώ στο ζήτημα το, όχι των απορριμμάτων. Είχα φέρει και φωτογραφίες σας δείξω σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει πλέον. Θα επικεντρωθώ στην οργή που υπάρχει στην Ευρώπη απέναντι σε, απέναντι σε, σε αυτά εδώ τα κάστρα που λειτουργούν σαν τα κάστρα του Κάφκα. Υπάρχει μια σιωπηλή οργή. Διαλέξατε σήμερα μεταξύ δικαίου και αδικίας, γιατί εμείς το καρβουνάρι, και θα μιλήσω για το καρβουνάρι, νιώθουμε μεγάλη αδικία, γιατί η καταστροφή είναι τεράστια. Την είδατε με τα μάτια σας και η ατιμορρησία, η ατιμορρησία όσων δημιούργησαν αυτή την καταστροφή και συνυπεύθυνοι αυτής της καταστροφής κατά εμέ είναι και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η ατιμορρησία θα μείνει όπως έχει και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα και θα δημιουργήσει, είναι ένα από αυτά τα μικρά προβλήματα που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις επόμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ την, την Επιτροπή σας για το ταξίδι που έκανε, αλλά για τη μορισία θα παραμείνει. Και αυτό είναι το λυπητερό σε αυτήν την ιστορία. Σας ευχαριστώ. Ε. Λοιπόν που δεν μπορείτε να καλυφθείτε από τον χρόνο που σας διαθέτουμε, αλλά έτσι κι ε, είναι έξτρα αυτός ο χρόνος, εκτός ημερησίας ε, διατάξεως. Και εκτός από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης σας δίνω και σας το λόγο κάτι το οποίο δεν προβλέπετε. Οπότε λυπούμε που ε, δεν καλυφθήκατε. Βεβαίω πρέπει να βλέπουμε το λόγο για τα μέλη τη Επιτροπή. Κύριε Χουντή. Ένα λεπτό και εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ειλικρινά δεν αντιλαμβάνουμε πώς έχει η διαδικασία τώρα. Αυτά που υπόθηκαν από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου και τις παρατηρήσεις των κυρίων Γκίκα και Παπαδόπουλου έπρεπε να τις είχαμε ακούσει κατά τη γνώμη μου πριν ψηφίσουμε. Τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό που κάνουμε. Το δέχομαι, είναι μια δημοκρατική ευαισθησία της Επιτροπής μας, αλλά Φαντάζομαι ότι αυτά που υπόθηκαν είτε από τον κύριο εκπρόσωπο του Υπουργείου είτε από του άλλου κύριου θα ελαμβάνονται υπόψη κατά την ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει έγιναν ό,τι έγιναν, αυτή είναι η έκθεσή μα, έχει πολλά θετικά στοιχεία. Εγώ απλώ θέλω να σα πω κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι που δεν ψηφίσατε την προφορική τροπολογία και ξέρετε ότι σε τέτοιε περιπτώσει αναλαμβάνουμε και εμεί ευθύνη. Τι έλεγε η προφορική τροπολογία για το γραμματικό, να γίνουν γεωτρήσει. Έχουμε πάμπολα παραδείγματα. Αναφέρομαι τελευταία μαυροράκι, σας το ανέφερα στη συζήτηση που κάναμε, κατάρρευση στη Σάμο, που οφείλεται ότι οι μελέτες δεν έγιναν με τα κατάλληλα τεχνικά όργανα ή δεν έγιναν ολοκληρωμένες. Με συνέπεια μετά το κόστος να είναι πολλαπλάσιο. Εδώ λοιπόν αν υιοθετούνταν η πρόταση, βεβαίως είναι στο χέρι του Υπουργείου, στο χέρι των ε, αρχών, οι κάτοικοι έχουν προσφερθεί με δικά του έξοδα να κάνουν αυτή επιτέλου τη γεώτρηση, να δουν που βρίσκεται ο υδροφόρο ορίζοντα και αν υπάρχει κίνδυνο για την υγεία και για όλη αυτή την υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να έχει εγγυηθεί κάποιο ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Διαφορετικά είναι επικίνδυνο για την υγεία. Ελπίζω να μην το βρούμε μπροστά μα. Διότι τότε πραγματικά θα έχουμε κλείσει τα μάτια μα σε κάτι πρόδειλο, σε κάτι αυτονόητο. Εν πάση περιπτώσει, α ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε διαφορετικά διότι δεν θέλω να αντιλέξω σε όσα είπε ο κύριος του, εκπρόσωπος του Υπουργείου, το σέβομαι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις αν πράγματι αυτά πραγματοποιούνται και αν είναι η σωστή μέθοδος. Ευχαριστώ για να μην φάω το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χούντι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν γνώμη ω προ την ψηφοφορία οι συνάδελφοι ένα λεπτό μόλι πριν από την ψηφοφορία. Δεν θα ήταν σωστό να ξανανοίξουμε το πεδίο ένα λεπτό πριν από την ψηφοφορία και γι' αυτό και ψηφίσαμε και νομίζω ότι με υπεύθυνο τρόπο ε, αξιολόγησαν την υπόθεση οι συνάδελφοι. Βέβαια θελήσαμε να ακούσουμε και τις διαφορετικές ούτως υπήν απόψεις των εκπροσώπων των πολιτών. Δεν πιστεύω όμως ότι θα μπορούσε αυτό να έχει επίδραση στην διεξαγωγή, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο κύριος Στουργάης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όπως είπατε, ε, τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει, να μην ανοίξουμε τώρα άλλη κουβέντα. Επισκεφθήκαμε επί τόπου την περιοχή και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλοι όσοι συμμετέσχομαι εκεί και η γραμματεία ε, άλλωστε εγκρίθηκε ομόφωνα η έκθεση από την Επιτροπή μας και θα πρέπει προς τις ελληνικές αρχές και προς τους ε, τον να τους πω ότι αυτό για μας είναι χάρτης πορείας. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε, να συνεργαζόμαστε. Νομίζω ότι υπήρξε καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση διακρίνεται από ισόρροπη δίκαιη αντιμετώπιση. Δεν έχω τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους και τους Έλληνες συναδέλφους που μας ε, βοήθησαν καθ' όλη αυτή την ε, αποστολή στο έργο μας και πάλι ευχαριστούμε. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε εσάς, εμείς κύριε Ιτουργκάτ και τον Υπουργό του Υπουργείου και τους Έλληνες Πολίτες και πάμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε τώρα την ε, έκθεση της κυρίας Ρετζίνα Σλάχ την 1690 του 12. Της δώσουμε το λόγο για 5 λεπτά για να μας ε, εξηγήσει ε, την εκθεσή της, την αναφορά της που αφορά την κατάρτιση των σας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω προσωπικό στο αίτημα αυτό, την αναφορά αυτή, ενώπιον της επιτροπής σα Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι για διάφορους λόγους παίρνουν το δρόμο της Ευρώπης και προσπαθούν να βρουν εδώ προστασία από πόλεμο και άλλους κινδύνους που αντιμετωπίζουν πολλές φορές και τι θα τα πω ότι γενικά θεωρείται, οι άνθρωποι αυτοί έχουν υψηλή κατάρτιση, αλλά δεν μπορούν να πάρουν τα πτυχία τους και τα διπλώματά τους μέσα σε αποσκευές τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε άσυλο ε, εάν και εφόσον τους δοθεί άδεια να εργαστούν, συνήθως απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες ή εποχιακές εργασίες. Πλην όμως μπορούν να περάσουν πολλά χρόνια για να μπορέσει ένα ετών το άσυλο να ε, νομιμοποιήσει την κατάστασή του ε, και μπορεί να μείνει για αρκετά χρόνια εδώ. Έτσι λοιπόν ε, χάνουν οι αιτούντες το άσυλο από την μακρόχρονη αυτή αναμονή την επικοινωνία, την επαφή με το επάγγελμά τους, την ικανότητα ακόμη και να το ασκήσουν. Έχουν όμως δικαίωμα στην εργασία και οι αιτούντες στο άσυλο. Και αν τους επιτρέψουμε να εργαστούν στο επάγγελμα το οποίο έχουν ε, μάθει, ε, προκύπτουν πάρα πολλές θετικές πτυχές για όλους τους εμπλεκόμενους, πιστεύουμε. Αυτό απαιτεί ωστόσο μια διαδικασία επαλήθευσης των ε, δεξιοτήτων, πρακτική και θεωρητική εξέταση ενδεχομένως και με υποστήριξη ως προς την διεξαγωγή αυτής της εξέτασης με βοήθεια δηλαδή, ε, ώστε να βεβαιωθεί ότι πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εξάσκηση ενός επαγγέλματος και βέβαια όταν αναγνωριστεί η δεξιότητα για την εξάσκηση ενός επαγγέλματος θα πρέπει αυτή να είναι αναγνωρισμένη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα λοιπόν να υπογραμμίσω ορισμένες θετικές πτυχές. Εάν επιτρέψουμε στους στο άσυλο να εργαστούν στο επάγγελμα που έχουν ε, μάθει, θα πρέπει να καταβάλλεται ο προβλεπόμενος από τον νόμο μισθός και έτσι δεν θα επιτρέπεται το κοινωνικό dumping ή το dumping ως προς τους μισθούς. Θα μπορούν να καταβάλουν τις εισφορές τους στο σύστημα ε, στο, κρατικό, στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Θα μπορούν να εξασφαλίσουν το βιοπορισμό τους και δεν θα είναι πια επέτες. Θα μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν ε, τα τραύματα, τις τραυμικές εμπειρίες του παρελθόντος η αγοραστική τους δύναμη θα αυξηθεί. Θα μπορούν να ε, εξασφαλίζουν αγαθά που δεν θα είναι μόνο τα βασικά αγαθά. Επίσης θα μπορούν να θα καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα, η μαύρη εργασία, η ανάπτυξη παράλληλων κοινωνιών και άρα μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα μια δυνατότητα εξίσωσης του αντιμετώπισης των προβλημάτων σε εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή αγορά και βεβαίως πιστεύω ότι θα υπάρχει θετική, θετικός αντίκτυπος και σε περίπτωση επανόδου του ετούντος του άσυλο στην ε, πατρίδα του γιατί και δεν θα έχει χάσει την επαφή με ε, το επάγγελμά του και θα έχει οικονομικά και κοινωνικά καλύτερες συνθήκες στην επιστροφή, στην χώρα προελεύσεως και ενδεχομένως θα έχει εξοικονομήσει, θα έχει αποταμιεύσει κάποια χρήματα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει στην χώρα προελεύσεως του. Έτσι λοιπόν η Ένωση Γυναικών Λουθυρανικών Εκκλησιών της Αυστρίας ζητά την ε, εξασφάλιση της δυνατότητας για τους ιστοτούντες στο άσυλο να εξασκούν το επάγγελμά τους, το επάγγελμα που έχουν μάθει, ή να ε, εντάσσονται σε ένα νέο επάγγελμα, να καταρτίζονται δηλαδή σε ένα νέο επάγγελμα και να μην χάνουν αυτή τη δυνατότητα για ε, εργασία και αξιοπρεπή ζωή. Ελπίζω να βρω υποστήριξη στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτής της αναφοράς. Παρακαλώ εκ μέρους της Επιτροπής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνούμε 100% με την ε, υπόβαλωση στην αναφορά σε σχέση με το κατά πόσον ε, είναι δυνατόν να εκμεταλλευτούμε τις δεξιότητες αυτών για τον άσυλο να αναγνωριστούν οι δεξιότητε τους και όπως είπαμε σε απάντησή μα, αυτά όλα διέπονται από την οδηγία του 2005 που ρυθμίζεται τη αναγνώριση των δεξιοτήτων που έχουν αποκριθεί στην Ευρώπη. Επίση, έχουμε και κάποιε άλλε διατάξει που αφορούν την αναγνώριση ε, των δεξιοτήτων που κανεί θέλει να αναγνωριστούν από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Αυτό ε, ισχύει για πολλέ κατηγορίε ε, ή θα γίνουν τρίτων χωρών, όπω και των ετών άσυλων και των προσφύγων. Οπότε θα πρέπει και εδώ πέρα να εφαρμοστεί αυτή τη μεταχείριση και ιδίω για του ετούντε άσυλο σα προτείνουμε και προσθέτουμε ότι πάρα πολλά έχουν αλλάξει από τότε που υπευλήθη η αναφορά, διότι στο μεταξύ έχουμε μια καινούργια δέσμη ρυθμίσεων για το άσυλο και έχουμε δύο οδηγίε που είναι πάρα πολύ σχετικέ Μία που αφορά του ε, ετούντε άσυλο, που επιτρέπει στου ετούντε άσυλο να ενταχθούν μετά από 9 και όχι 12 μήνε στην αγορά εργασία. Και έτσι καλύπτονται αυτά τα οποία ζητεί ε, η αναφορά Και έτσι δεν θα έχουμε αυτή την κατασπατάληση του ανθρωπίνου δυναμικού, γιατί θα μπορούν να κάνουν την τέχνη του ούτως επί αυτοί οι άνθρωποι. Η δεύτερη είναι η οδηγία για τις ε, δεξιότητες που και αυτή καλύπτει αυτό το οποίο ζητεί αναφορά και λέει για τους επιμετές άσυλο που έρχονται εδώ, δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν έχουν έγγραφα να αποδεικνύουν τις δεξιότητές τους. Οπότε ε, αυτό γίνεται γιατί πολλοί φορέ άνθρωποι πρέπει να φύγουν βιαστικά, γιατί απειλεί το η ζωή του από τη χώρα του. Και έτσι να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην διεθνή αυτή προστασία και έτσι έχουμε εξαιρετική ε, μεταχείριση σε σχέση με τη συνήθεια διαδικασία για αναγνώριση των δεξιοτήτων. Τα κρατημέλη θα πρέπει να, να δεχτούν και να ρυθμίσουν αντίστοιχα στην νομοθεσία τους αυτές τις ρυθμίσεις και προβλέπονται και κάποια νίκη στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη με αυτή την αναγνώριση των δεξιοτήτων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μπέκερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ θα ήθελα εν συντομία να συνοψίσω το πώς ε, κρίνω εγώ αυτή την ε, αναφορά. Καταρχάς καλωσορίζω τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως αυτές που μας ε, περιεγράφησαν μόλις τώρα, τις τελευταίες δραστηριότητες, οι οποίες δείχνουν ότι είναι σωστή η κατεύθυνση και άρα βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία αρμοδιότητα με μια αρχή και μόνο που θα πρέπει να πιστεί. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των δικών τους νομοθετικών αρμοδιοτήτων θα πρέπει να προσδιορίσουν φερρυπίν τις προθεσμίες, πόσο, καιρό θα πρέπει να έχει περάσει, καιρός θα πρέπει να έχει περάσει πριν ζητήσει τη δυνατότητα για πρόσβαση στην αγορά εργασία ο ετών το άσυλο. Αυτά τα πράγματα θα τα ρυθμίσουν τα κράτη-μέλη. Πάντως ένα-δύο πράγματα που θα μπορούσαμε εμείς ως Επιτροπή να μελετήσουμε θα ήταν καταρχάς το ενδεχόμενο αυτή η αναφορά να παραπενθεί σε επιτροπές πολιτικών ελευθεριών και απασχόλησης παράλληλα με το σχολιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ζητήσουμε την περαιτέρω επεξεργασία της. Και δεύτερον, με μια προφορική ερώτηση oral inquiry προς το Συμβούλιο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την ε, τοποθέτηση των κρατών μελών για την κάθε περίπτωση, για το κάθε κράτος μέλος χωριστά δηλαδή, σε σχέση με τους ετούντες στο άσυλο και τις προτάσεις που διατυπώνονται εδώ. Δηλαδή τη δυνατότητα για επαλήθευση επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα μπορούσε να οργανωθεί. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και να ζητήσουμε από το Συμβούλιο τις απαντήσεις. Και νομίζω ότι έχουμε περιθώριο ακόμη στη διάρκεια της τρέχουσα θητεία του Κοινοβουλίου να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Νομίζω ότι στο θέμα αυτό έχει η Επιτροπή απαντήσει με μια με ένα έγγραφο το οποίο ασφαλώς αναφέρεται στην υπόθεση αυτή, μελετάει την υπόθεση αυτή και ίσως μπορεί και στη διαδικασία την νομοθετική να ενταχθεί. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι μέχρι, μέσα σε μια-δυο μέρες θα έχει λυθεί το θέμα, αλλά πάντως αποτελεί καλό ε, ιονό. Η προσπάθεια επίσης για επιτάχυνση των διαδικασιών για τη χορήγηση απάντησης στο αίτημα του κυρίου Μπέκερ, την οποία τυπικός βέβαια υποστηρίζω, αλλά επί της ουσίας δεν νομίζω ότι θα ευοδοθεί, γιατί κλείνει πράγματι, τελειώνει πια η θητεία μας και ήδη εδώ και κάποιους μήνες η Προεδρία του Συμβουλίου δεν ε, εγγράφει στις ημερήσιες διατάξεις των εργασιών τις δικές μας προτάσεις, αλλά και άλλων επιτροπών, γιατί έχει άλλα κατεπήγοντα ζητήματα που εγγράφει για τις ε, συνόδους ολομέλειας. Έτσι λοιπόν, ίσως θα μπορούσε ο κύριος Μπέκερ αυτό το θέμα να το υποβάλει για συζήτηση στους συντονιστές, προκειμένου να ληφθεί απόφαση και να μείνει ανοιχτή η αναφορά, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε, παράλληλα βέβαια και με την Επιτροπή που μας υπόσχεται ότι θα παρακολουθήσει την υπόθεση, την εξέλιξή της με τη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ την αναφερόμενη που το ζήτησε και κλείνω προς το παρόν τη συζήτηση στο θέμα αυτό και περνάω στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης αναφορά της κυρίας Πουλπάν σχετικά με τη συμμετοχή σε Αθλητικού αγώνε και λοιπέ αθλητικέ εκδηλώσει μεταναστών που δεν έχουν την ηθαγένεια μια Ευρωπαϊκή Χώρα. Ο κύριος η κυρία Ρενάτα Μοναστέρο είναι εδώ και παρακαλώ να μα κάνει την παρουσίαση. Πριν όμως από αυτό έχουμε ένα βίντεο να δούμε. Όχι, όχι, πρώτα λαμβάνει το λόγο και μετά συζητάμε. Βλέπουμε το βίντεο. Καλημέρα Πρόεδρε Ματζόνη και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καλημέρα και προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι εδώ ως εκπρόσωπος της ΦΙΛΣΕΜ, που είναι η, Ιταλική Ομοσπονδία των Αλλοδαπών στην Ευρώπη και, στον, και στην Μεσόγειο. Θα σας παρουσιάσω αυτή την αναφορά που αφορά τα, τους ανηλίκους οι οποίοι φυσικά διακρίσεις στα σπορ και έχουμε πληγεί από τέτοιε μηνύ διακρίσει και γι' αυτό και κάναμε αυτό τον φορέα στη Νάπολη και τίποτα δεν άλλαξε όμω. Οπότε και στράφημε προ ε, τη δική σα επιτροπή. Θεωρούμε ότι αυτό είναι η τελευταία ευκαιρία, ούτω ώστε κάτι να γίνει για να ε, λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Και με την άδεια σας θα παρουσιάσω αυτό το, το, το, το, το βίντεο που αφορά την αναφορά μας. Ε, senza audio. Χωρίς ήχο, λέει ο πρόεδρος. Έχουν τους τίτλους, έχουν μεταφραστεί. Αν θέλετε διαβάζω. Se può ripassare l'immagine. Sono tutti titoli di Πρόκειται για τίτλους εφημερίδων. sport e cittadinanza Il sogno azzurro di Daria, nata in Ucraina ma da 11 anni in Italia, per un documento non... Το όνειρο της ε, Δαρίας που γεννήθηκε στην Ουκρανία, αλλά επειδή δεν έχει ε, τα σχετικά έγγραφα, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές εκδηλώσεις. Okay. Promessa sincro non può gareggiare perché straniera, niente tuffi per ragazzina di 10 anni. Συγχρονισμένη κολύμβηση και καταδύσεις. Ε, εκεί έχουμε κάποιον στην Πάντοβα αφρικανική καταγωγή που δεν μπορεί να συμμετάσχει ακριβώ γιατί είναι αλλοδαπτή. Επίση έχουμε την Νάντια Σβήτρη. Είναι μαροκινής καταγωγή και δεν μπορεί να συμμετάσχει στους αγώνες στην Ταϊβάν όσον αφορά το πατινάζ ε, και περιμένει την ηθαγένεια τέσσερα χρόνια. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Onorgoglio διέστερε essere cittadina Ρωμίνα. Δεν ακούγεται καλά η ομιλήτρια γιατί είναι μακριά από το μικρόφωνο. Punto il dito verso i regolamenti sportivi e non verso l'Italia che è un paese meraviglioso. Το βίντεο δεν ακούγεται καλά και δεν μπορεί να μεταφραστεί. Unire e non separare. Lo sport è cultura, uguaglianza e gioco per tutti i bambini del mondo. L'unione και έχουμε τώρα αυτή την προσπάθεια για άνοδο της ποιότητας των αθλητισμών. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο καταπολεμεί την ε, δυσμενή διάκριση, και αυτό θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ο αθλητισμός επομένως για να μπορέσει να ωφεληθεί με τη σειρά του θα πρέπει να σταματήσει να υποβοηθά τις δυσμενείς διακρίση θα πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φραγμοί το, το, το, το, το πλήρες δικαίωμα συμμετοχή όλων και κυρίως όσον αφορά του ανηλίκου. Όλοι οι ανηλίκοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτω καταγωγή και ηθαγένεια. Και θα πρέπει αυτό να ισχύει για όλα τα επίπεδα και θα πρέπει να είναι δυνατόν να συμμετέχουν ελεύθερα όπου επιλέγουν, σε όποια χώρα επιλέγουν ή στη χώρα που μένουν οι ανήλικοι. Άρα αυτό θα πρέπει να το καταφέρουμε και αυτό θα πρέπει να γίνει με πράξεις, όχι μόνο με λόγια. Ξεκίνησαμε αυτή την προσπάθεια εμείς, αλλά τώρα από εσά εξαρτάται για να μας βοηθήσετε να πετύχουμε το στόχο μας. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Βρίσκουμε και την κυρία Πούλπαν για αυτό το βίντεο. Ζανλούκα Μόντα για την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι συμφωνούμε με αυτήν την αναφορά. Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ε, ως εξής. Πρώτα-πρώτα, από πλευρά νομικής, τονίζουμε ότι τις δυσμενείς διακρίσεις βάσει της ταγένειας απαγορεύουν τη δύναμη του άρθρου 18 της συνθήκης και αυτό ισχύει και για τον αθλητισμό ρητά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, η σχέση ηθαγένειας και ε, αθλητισμού, υπήρχε το 2010, κατόπιν μιας μελέτης. Τα συμπεράσματα ήταν βασικά το ότι η πρόσβαση στην άσκηση του αθλητισμού και η συμμετοχή στους αγώνες σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ελεύθερη. Δεν θα πρέπει να πλήσετε από διακρίσεις βάσει της ηθαγένειας. Οι ενδεχόμενες δυσμενείς διακρίσεις θα πρέπει να είναι πάρα πολύ λίγες και πάρα πολύ συγκεκριμένες, όπως με το ΔΕΚ ε, έχει πει ότι υπάρχει περισμός όσον αφορά τις εθνικές ε, ομάδες ή την απονομή κάποιων μεταλλίων. Αλλά θα πρέπει ο κανόνας να είναι ανοιχτή πρόσβαση. Αυτό από πλευράς νομικής. Αλλω μπορεί να έχουμε διαδικασία παραβάση, ούτω ώστε να αρθεί η τυχόν ε, δυσμενή διάκριση. Τώρα άλλη απάντηση από άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε σε σχέση με την αναφορά αυτή ότι ο, το, τόσο ο αθλητισμός όντως είναι τρόπος ένταξης, συμμετοχή που μένω των πολιτών αυτό το έχει αναγνωρίσει σε μια σειρά εγγράφων το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε μια ανακοίνωση του 2011 όπως λέει και αναφορά και έχουμε επίσης και μια σειρά ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου έκθεση ε, του κ. Μαυρομάτη και κάποια άλλη έκθεση, κάποιο άλλο ψήφισμα του Κοινοβουλίου και επίσης το 2014 επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Erasmus Συν, το Erasmus Plus ε, που έχει έναν ε, κεφάλαιο για τον αθλητισμό και ο στόχος είναι η καταπολέμηση ε, του ρατσισμού, των σημερινών διακρίσεων μέσω του αθλητισμού όλα αυτά και θα πρέπει μέσα αυτό να το, να το εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, οι αθλητικές ενώσεις και αυτός του στόχος να προάγουν. Σας ευχαριστώ, Μελή Πρόεδρος πάρα πολύ θετικά αυτά τα οποία λέτε. Θέλει κάποιο συνάδελφο το λόγο για αυτό το θέμα. Δεν ζητεί κανείς το λόγο. Οπότε, με δεδομένη απάντηση της ε, Επιτροπή, θα μείνει ανοιχτή μια αναφορά. Και επομένως, αν θέλουν οι ετούντες, μπορούν να προσθέσουν κάτι και να δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφύγει στο δικαστήριο επί παραβάση κατά της Ιταλίας. Οπότε σε... θα δούμε τι θέλουν τυχόν να προσθέσουν οι υποβάλλοντες αναφορά και ενδεχομένω αυτό ο φορέα ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιου πόρου που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέτοιε περιπτώσει. Σα ευχαριστούμε κυρία Πούλπαν για την ε, αναφορά και όμως κλείνουμε αυτό το σημείο της διάταξης και προχωρούμε στο επόμενο. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Παλιαδέλη, την αντιπρόεδρο, η οποία πρόκειται να με αντικαταστήσει όσον αφορά τη διεξαγωγή των εργασιών μα. So, let's have five minutes break. Κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, λέει η κυρία Παλιαδέλη, για να έρθουν οι υποβαρόντες στην αναφορά.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 Εγώ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

Um, θα έπρεπε να έχουμε αρχίσει πριν από πέντε λεπτά, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για το θέμα και γι' αυτό θα περιμένουμε την άφηξή τους από στιγμή σε στιγμή. Αν θέλετε να αρχίσω τώρα, αρχίζω. Θέλετε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα. Σημείο 20 του κυρίου Βιντσέντσο Αντωνούτσο. Αρχίστε. Μάλιστα. Υποβάλλω μια αναφορά για την περίπτωση των δύο θυγατέρων μου και θα σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση από τις 17 Οκτωβρίου που έκανα την πρώτη παρουσίαση τις τελευταίες εξελίξεις. Όλα όσα θα σας πω είναι τεκμηριωμένα, δηλαδή επειδή σε τρία λεπτά δεν μπορώ να σας δείξω όλα τα έγγραφα, μπορώ όμως αν ενδιαφέρεστε να σας τα υποβάλω. Δυστυχώς ο υπολογιστής δεν δουλεύει, αλλά εγώ δεν μπορώ να δω ελεύθερα τις κόρες μου από τον Μάιο του 8 από την τελευταία ψηφοφορία στις 17 Οκτωβρίου εδώ σε αυτή την Επιτροπή έλαβα μόνον τρεις ανακοινώσεις από τις δανέζικες αρχές δηλαδή τρία αιτήματα πληρωμής διατροφής τα οποία και έκανα. Για όλα τα υπόλοιπα δεν έλαβα καμία πληροφόρηση. Συνεχίζω να μην μου, ε, ε, συνεχίζουν να μην μου επιτρέπουν επαφές άμεσες με τις κόρες μου. Έχω επισκεπτικά δικαιώματα, αλλά δεν μπορώ να πάω στη Δανία για να δω τις κόρες μου. γιατί η μητέρα ελέγχει όλες τις επαφές. Όσο για τις δανέζικες αρχές, όταν ζητώ έρευνα για την περίπτωση, απάντησαν πριν από πολύ καιρό ότι δεν έχουν αρκετά εκπαιδευμένο προσωπικό για να μπορέσουν να ερευνήσουν την περίπτωσή μου. Το μόνο που θέλω να σας πω εδώ, σε αυτό το πολύ λίγο χρόνο που διαθέτω, είναι ότι πρέπει να σκεφτείτε ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχει και η δική μου περίπτωση και άλλων αναφερομένων ή αναφερόντων, ότι δεν υπάρχει συνεχής επαφή πια μεταξύ γονέων και παιδιών. Είναι γνωστό ότι όταν καταστρέφεται μια επαφή μεταξύ ενός γονέα και του παιδιού, ιδίω αν είναι κάτω των 10 ετών το παιδί, είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, στο μέλλον να έχει κανείς κανονικές επαφές. Θεωρώ λοιπόν ότι η Δανία παραβιάζει διάφορα άρθρα συμβάσεων του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, ιδιαίτερα ένα που είναι το 12, δεν μπορώ να σας το δείξω δυστυχώ, αλλά το έχω στην παρουσίασή μου και επίσης παραβιάζει το άρθρο 21.3 της Συνθήκης της Χάγης που έχει υπογράψει η Δανία και τις δύο. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι μια έκκληση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να παρετηθείτε από την περίπτωση αυτή γιατί τα μαθήματα που πήραν οι κόρες μου είναι ότι α ναι, α, ναι, ναι. Ναι, αν έχω λίγο χρόνο μπορώ να τα... Όχι αυτό, είναι ένα έγγραφο PDF. δεν το δείχνει. το δεξί βέλος προχωράει, όχι με το κάτω. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι στη συνθήκη για τα δικαιώματα των παιδιών του ΟΗΕ υπάρχει το δικαίωμα σε τακτική βάση να βλέπουν τους γονείς τους σε άμεσες συναντήσεις. Επομένως συμπερασματικά τα παιδιά μας θα είναι οι αυριανοί Ευρωπαίοι αν αυτές οι επανειλημμένες παραβιάσεις βασικών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνουν αποδεκτές στην Ευρώπη ανεκτές, τότε δεν καταλαβαίνω τι είδους Ευρωπαίος πολίτης θα μεγαλώσει. Ευχαριστώ. Εκπροσωπείτε και άλλους δύο αναφέροντες. Ναι, μάλιστα. Για τον Φαμπρίτσιο Ινφάντε, μάλιστα. Λοιπόν, ο Φαβρίκιος δεν έχει και αυτός δικαιώματα επίσκεψης της κόρης του Μαρτίνα Ινφάντε. Κανένα, καμία Δανέζικη Ευρωπαϊκή Αρχή δεν με έχει πληροφορήσει εδώ και πάνω από 11 χρόνια δεν έχω νέα για τη Μαρτίνα. Είναι απαράδεκτη και βάρβαρη συμπεριφορά προς έναν πατέρα και την κόρη του. Κατά τα χρόνια αυτά η Δανία δεν προσπάθησε παρά μόνο να αποφύγει επαφές με μένα. Έμαθα ότι άλλαξε και το επίθετό της χωρίς τη συγκατάθεσή μου και ότι στη Δανία έχει ξαναβαπτιστεί παρά το ότι είχε βαπτιστεί ήδη στην Ιταλία. Και τα ψέματα έφτασαν σε τέτοιο σημείο ώστε μου είπαν ότι μόνο όταν θα γίνει 18 χρονών θα μπορέσω να τη δω. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Φαβρικίου Ινφάντε. Και για τον επόμενο αναφέροντα. Ναι, ορίστε η δήλωση του Κεν Κούπερ. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών, στις 12 Δεκεμβρίου 2013 έμαθα ότι η Δανέζικη κυβέρνηση μυστικά κρατούσε στοιχεία για τα email μου και τις διαλέξεις μου παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα μου. Μου λένε ότι η Δανέζικη κυβέρνηση έχει κάνει παρόμοιες παρακολουθήσεις και για άλλους αναφέροντες. Ένας από αυτούς έχει δει και στοιχεία της παρακολούθησης του με τα μάτια του. Καταγεγραμμένες διαλέξεις ας πούμε. Η γραμματεία έχει λεπτομέρειες για τα έγγραφα αυτά και που μπορεί κανείς να τα βρει. Λυπάμαι, αλλά δεν δουλεύει πάλι το ρημάδι. Α, να το διαβάσω. Α, ναι, ναι. Ζητώ από την Επιτροπή σας επίσημα να ζητήσει από την κυρία Χέλε Τόρνινγκ Σμιτ, Πρωθυπουργό της Δανίας, αντίγραφα όλων των εγγράφων που αφορούν κυβερνητική κατασκοπία εναντίον μου και οποιοδήποτε άλλο αναφέροντος. Επίση ζητώ η Επιτροπή να κάνει δύο πρόσθετα πράγματα Πρώτον ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις κατά της Δανία σε ύψο 500 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον. Η Ένωση έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέτοια πρόστιμα όπως το έχει ξανακάνει γιατί οι περιπτώσεις μας δικαιολογούν τέτοια οικονομι... τέτοιες οικονομικές κυρώσεις. Δεύτερον, ζητώ από την Επιτροπή σας να υποβάλλετε εξ ονόματός σας αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα συνεργαστώ με τα χαράς μαζί σας για αυτό το θέμα. Η Γραμματεία επίσης έχει έγγραφα για όλες τις προσπάθειές μας σχετικώς. Τέλος παρακαλώ να καταλάβετε ότι οι αναφορές μας δεν αφορούν απλώς μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις κυδαιμονίας όπως λέει η Βιδανέζικη κυβέρνηση. Όχι, οι αναφορές μας αφορούν ένα, μια συστηματική παραβίαση και διαφθορά της κυβέρνησης. Παραδείγματο χάρη, κυβερνητικοί αξιωματούχοι που επανειλημμένως μας λένε ψέματα συνεργάζονται για να πάρουν τα δικαστήρια αποφάσεις εναντίον μας. Αγνοούν, βασικά στοιχεία, επιλεκτικά εφαρμόζουν τον νόμο. Ε, τον εφαρμόζουν μόνο όταν ωφελεί δανούς γονείς και επιτίθενται επιθετικά κατά των δικηγόρων μας. Βάζουν ξένες μητέρες στη φυλακή, μας κατασκοπεύουν γιατί τολμήσαμε να έρθουμε μπροστά στην Επιτροπή σας. Όλα αυτά παράνομα μας αρνούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά μας απλώς γιατί δεν είμαστε δανείοι. Αυτές είναι σοβιετικές τακτικές. Δεν έχουν καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι παράνομες και ανήθικες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ματσόνη και όλη την Επιτροπή σας και σας παρακαλώ να δώσετε συνέχεια στο θέμα. Κέντ Κούπερ, 11 Φεβρουαρίου 2014. Εμείς σας ευχαριστούμε και να σας ενημερώσω συναδελφοί ότι πρόκειται να συζητήσουμε πρώτα τις αναφορές, οι θα κάνουν την εισήγησή τους και κατόπιν θα ακούσουμε ε, τη γνώμη της Επιτροπής. Στο τέλος. Πρώτα παρουσιάσει και μετά μιλήσει η Επιτροπή. Δεκαεπτά, δεκαεννέα και είκοσι τρία. Η κυρία Μάριον Βάιλχάρτερ. σας παρουσιάσω τη δεύτερη αναφορά μας σήμερα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτέ. ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη δεύτερη αναφορά μας. Πολλοί εξημών έχουν μπορέσει να μάθουν ποιες είναι αυτές οι συνέπειες αυτές της του αποχωρισμού με τα παιδιά και τις μη συμμόρφωση με τι ε, αποφάσει, γιατί πρόκειται εδώ πέρα για μια κατάφορα παραγωγή των δικαιωμάτων και για δυσμενή διάκριση την οποία έχουν διαπράξει οι αρχέ τη Δανία. Σύμφωνα ε, με, με το ΕΕ πρόκειται εδώ πέρα για κακομεταχείριση κατά του ανηλίκου. Πρόκειται περί απαγωγής οι ιδανικές αρχέ δεν συνεργάστηκαν. Παρά το ότι υπάρχει καταδίκη του πατέρα που απήγαγε το παιδί από τα ποινικά δικαστήρια, αρνούνται να βοηθήσουν. Πρόκειται για έγκλημα που έχει γίνει κατά του Φανιλίκου του Όλιβερ το 2010 ο Φρέντερ Κίλμπρο που είναι εμπειρογνώμος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τώρα πρόκειται να γίνει ε, ο δικαστής του τη Ιδανίας στο, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε το 2012 ότι ο Όλιβερ θα πρέπει να επιστρέψει σε μένα. Όμως οι νέες αρχές αγνώρισαν ε, αυτή την απόφαση του δικαστού. Επίσης έχουμε και απόφαση του ΟΗΕ που λέει ότι η Δανία θα πρέπει να μου επιτρέψει να βλέπω ε, το παιδί μου. Το αγνώρισαν και αυτό οι αρχές της Δανία η κυρία Άουκεν από παλιότερες περιπτώσεις ε, γνωριζόμαστε και γνωρίζει ότι εγώ δεν είμαι η εξαίρεση, δεν είμαι μοναδική τέτοια περίπτωση. Αν, αν κλείσετε τις αναφορές θα αποδείξετε ότι ο χάρτης των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι άκυρος. Ότι δεν ισχύει και ότι τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στερούνται δικαιωμάτων. Τέλος τελευταίο αλλά σημαντικό, θα πρέπει να σας διαβάσω ε, ένα κομμάτι από μια επιστολή που έλαβα τον Ιανουάριο από το Δανέζικο Υπουργείο Δικαιοσύνης όταν ξαναζήτησα να μου δώσουν κάποια στοιχεία σε σχέση με το παιδί μου. Επιλέξει, γράφει ότι σύμφωνα με 32 περί επισήμων γράφων το δικαίωμα στην πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί στον βαθμό που χρειάζεται ούτως ώστε να, να... Ε... να εφαρμόσουμε την ε, ασκούμενη πολιτική, την εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με διεθνή θεσμικά όργανα ή άλλες χώρες. Κατά τη γνώμη του Υπουργείου, εδώ υπάρχει επικείμενος ε, κίνδυνος και άμεσος κίνδυνος να διακυβευτούν τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής της Δανίας εάν αυτά τα έγγραφα και οι σχετικές πληροφορίες δημοσιοποιηθούν. Το Υπουργείο εστάθμιζε το κατά πόσο θα πρέπει αυτές τις πληροφορίες να δημοσιοποιηθούν και έκρινε κατά αξιολογήσεως και αφού εστάθμισε και τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής Δανίας ότι αυτά τα συμφέροντα κατησχύουν και επομένω δεν μπόρεσε να μου δώσει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Θα σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Παρακαλώ, βοηθήστε όλα αυτά τα παιδιά που περιμένουν πώς και πώς τη βοήθειά σας. Η Πρόεδρος, θέλετε να συνεχίσετε με τις επόμενες δύο αναφορές. Έχουμε τώρα την αναφορά που αφορά κάποια Αμερικανίδα μητέρα. Λέγεται Kim, Και μπορώ να σας δείξω ένα βίντεο το οποίο μας έχει στείλει. Η κύμα Μουσολίν. Does she know My name is Ονομάζομαι Κίμα Σπίνη Μουσολίνη και είμαι Αμερικανίδα. Έζησα στη Δανία το 1997 και 2012. Ε, ο γιο μου ονομάζεται Κόντι Κέντ Γιώχανσεν. Ε, έχει την ιθαγία την Αμερικανική και την Δανέζικη και αναγκάστηκε να μείνει στη Δανία με τον πρώην σύζυγό μου, τον Χένρι Γιώχανσεν. Από τον Νοέμβριο του 2012. Τον Αύγουστο του 2007 ε, ο πατέρα μου έπαθε καρκίνο και του είπαν ότι δεν θα ζήσει πολύ. Πέρασα τρει μήνε με τον πατέρα μου για να τον βοηθήσω και να τον αποχαιρετήσω. Ο Χένικ δεν επέτρεψε στον Κόντι να έρθει μαζί μου και να επισκεφτεί τον παππού του που πέθανε, οπότε και εγώ τηλεφωνούσα κάθε εβδομάδα για να μιλήσω τον Κόντι ε, από την Αμερική στη Δανία. Τον Οκτώβριο, πριν γυρίσω στη Δανία, προσπάθησα να, έχω, να, πετύχω την ε, γονική ε, μου να την μοιραστώ με τον πατέρα μου και μου είπαν ότι ξεκινάει τότε η, η διαδικασία για αυτό αλλά όμως χωρίς να το ξέρω πέτυχε ο πρασιζικός μου να έχει μόνο αυτό στη γονική παροχή και ε, τότε προς έκπληξή μου οι αρχές και τα για δικαστήρια έδωσαν τη γονική μέρημνα στον πρώην σύζυγό μου γιατί μου είπαν ότι είμαι αλλοδαπή. Αλλά δεν υπήρχε λόγο να μου φέρουν τη γονική μέρημνα. Πάντοτε ήμουν πάρα πολύ καλή μάνα και θέλει να είναι σε επαφή μαζί μου ο γιος μου, δεν είμαι βίαιη, δεν χρησιμοποιώ ναρκωτικά, ούτε είμαι αλκοολική, ούτε έχω κάποιο είδους ψυχολογική αστάθεια τον εμποδίζουν να με επισκεφθεί, ούτε καν δεν τον αφήνουν να χρησιμοποιήσει τηλέφωνο ή το Skype και οι αρχές της χώρας δεν εφαρμόζουν ε, τα, τις του δικαστηρίου για το δικαίωμα επίσκεψης και ε, έχω την έγγραφη διαβεβαίωση από το πεδίο ότι ε, το, τα έχει πει αυτά στους δασκάλους του, έχει τραυματιστεί ψυχολογικά από αυτό και τέλος πάντων όλα αυτά αφορούν το ότι δεν έχω την η ηθαγένεια διότι στη χώρα εκείνη δεν αναγνωρίζω τα δικαιώματα ε, μιας τέτοιας ε, ε, Έτσι είναι το σύστημα εκεί άσχετα με το τι ψέματα μπορεί να πει κάποιος ε, δανός. Ζητώ να πάρει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κατάσταση αυτή είναι αφόρητη. Ε, έτσι έχουν πληγεί πάρα πολλοί αλλοδαποί γονείς και τα παιδιά τους στην Δανία. Αφορά ο, ο κάθε στρώμα της δανεικής κοινωνίας. Ούτε το νομικό σύστημα στη Δανία παρέχει κάποιο ένδικα μέσα. Παρακαλώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μου αποδώσει πάλι τα δικαιώματα που έχω στην οικογενειακή ζωή σε σχέση με το παιδί μου. Να έχω το δικαίωμα, να το δω. Γι' αυτό αφορά όλους τους αλλοδαπούς επομένως ε, ε γονείς που έχουν παιδιά με δανός. Και επειδή δεν είναι δανείοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όλα αυτά καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών. Θα πρέπει επίσης να επιτραπεί το να μπορούν να διαμείνουν ελεύθερα και μόνιμα στη χώρα οι αλλοδαποί ε, γονεί, αφού ε, τα παιδιά τους δεν επιτρέπεται να φύγουν από τη χώρα. Οι αλλοδαποί αυτοί να έχουν ε, νομική προστασία όσον αφορά τα παιδιά τους και να επιτρέπεται τελικά στα παιδιά αυτά να ταξιδέψουν εκτός Δανίας όπως επιτρέπεται να το κάνει κάθε Δανός. Παρακαλώ τώρα να κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προσφύγει στις ε, Δανεικές Αρχές ε, προς όφελος των ε, παιδιών και των αλλαδαπών γονέων τους. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων και των γονέων και των ανηλίκων που γίνεται στη Δανία. Η σας ενημερώνω το ότι αυτό ήταν ε, το 29, η αναφορά υπαρθμών 29. Πρέπει τώρα να επιστρέψουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ή 17. Παρακαλώ, συνεχίστε. Μια Αμερικανίδα. Επίσης, η Τάμι Νόργκερτ. Πάλι έχουμε τραγικές εξελίξεις στην υπόθεση. Το μόνο που μπορώ να σας δώσω είναι πληροφορίες γενικές για τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στη, στη γυναίκα αυτή, γυναίκα και μητέρα. Ξέρουμε ότι η κόρη της έχει φύγει αρκετές φορές από το σπίτι. Η μητέρα έχει φυλακιστεί. Της έχει αφαιρεθεί μάλλον το παιδί και ε, έχει φυλακιστεί με την ε, κατηγορία της απαγωγής. Όταν όμως έφευγε το παιδί, η μητέρα ήταν ήδη στη φυλακή. Η αστυνομία της Δανίας έλαβε και επιστολή από τη μία, την κόρη, ότι η μητέρα της δεν ήταν καν ενήμερη ότι φεύγει, ότι έφυγε από το σπίτι κρυφά με συγγνώμη που προξένει σε φασαρία κτλ. Και η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ότι από την αποφυλάκηση της μητέρας, λόγω όπως ονομάστηκαν τεχνικών σφαλμάτων σε περίοδο δικαστικής διαδικασίας, Πράγμα το οποίο αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά με. Γιατί όταν κάποιο έχει φυλακιστεί χωρί να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο ή και διερμηνέα, δεν μπορεί να είναι σωστό. Αποφυλακίστηκε λοιπόν μετά. Και από ό,τι μαθαίνω η κόρη έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο πατέρας έχει ξεκινήσει μία, ένα δικαστικό αγώνα για τη διεκδίκηση του παιδιού που έφυγε από το σπίτι. Και η μητέρα βρίσκεται σε μία κατάσταση στην οποία δεν ξέρει πώς να χειριστεί πια στέλνει ενημέρωση στην Επιτροπή σας με εξελίξεις, με τις τελευταίες εξελίξεις μόλις συμβεί κάτι πιο συγκεκριμένο. Καλώς λέει η πρόεδρος, παρακαλώ να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε. Για την κυρία Σπελίν. Έχουμε την κυρία Μαρία Σπελίν από τις Φιλιππίνες που με κάλεσε να σας διαβάσω την αναφορά της προς την Επιτροπή. Ελπίζουμε τον να μας υποστηρίξετε στην ε, υπόθεση τη σχετική με τη δικαστικό αγώνα που είχαμε στη Δανία το 2013. Ε, φυσικά ε, με το γιο μου επιλέγουμε που θα ζήσουμε. Πήγαμε στις Φιλιππίνες όπου είμαστε ασφαλείς. Θέλουμε την υποστήριξη των φίλων και των συγγενών μας. Έχουν περάσει δύο μήνες στη Δανία όπου στερήθηκα το γιο μου όπου δεν είχα σταθερή διαμονή, δεν είχα την άδεια να εργαστώ για το μεγαλύτερο διάστημα, όπου ήμουν αντιμέτωπη με ένα σύστημα το οποίο δεν με ρημνούσε για την ε, ευημερία, για το καλό του παιδιού μου, το οποίο με δοκίμασε σκληρά. Και οι συνέπειες αυτής της ε, κατάστασης μπορεί να φανούν πολύ αργότερα ακόμα. Βρήκα τυχαία στο σπίτι της πρώην πεθεράς μου ένα έγγραφο το οποίο έλεγε το παιδί ήταν ε, σε ένα παιδικό σταθμό. Και έτσι πήγα στον, ε, στο δημοτικό διαμέρισμα για να ενημερωθώ για την κατάσταση του παιδιού μου. Του είπα ότι δεν είχα δώσει την άδειά μου να πάει στο παιδικό σταθμό το παιδί αυτό, αλλά μου είπαν ότι δεν είχα εγώ δικαίωμα, ότι κάνω τον επισκεφθώ και ότι κάθε γονιό, δηλαδή ο Δανό πατέρα μπορούσε να το στείλει σε όποιο σταθμό θέλει. Και δεν ήθελα να δω το γιο μου, εφόσον συνεργαζόμουν με τον πατέρα του, θα μπορούσα να τον βλέπω δύο φορέ τη βδομάδα μέχρι τέσσερι ώρε το πολύ. Διαφορετικά θα τον βάζαν σε ανάδοχη οικογένεια. Αποφάσει που έλαβαν κάποιοι άνθρωποι με στόχο και μέρημνα την προστασία του άντρα μου, του δανού άντρα μου, πρώην άντρα μου και όχι του παιδιού μου. ούτε καν όταν διεκδίκησα ισότιμη πρόσβαση προς τους δύο γονείς για το παιδί μου δεν εισακούστηκα. Γιατί διαπίστωσαν εκεί ότι δεν είμαστε κάτοικοι Δανίας. Είχα την τύχη να βρω δικηγόρο, ο οποίος κανονικά δεν δεχόταν ε, τέτοιου είδους υποθέσεις, αλλά με δέχθηκε και η διαδικασία της, ε, η, δωρεάν αυτή διαδικασία με τη δικαστική αρρωγή την οποία δέχθηκε κατ' εξαίρεση ο δικηγόρος ε, δεν ήταν τόσο δωρεάν όσο φάνηκε αρχικά γιατί χρειάστηκε να πληρώσουμε πολλά λεφτά και η οικογένειά μου στις και εγώ. Όταν μπορέσαμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μου ε, δόθηκε η εντολή από το δικαστήριο μια φορά τη βδομάδα να παίρνει ο άντρας μου το παιδί μια φορά κάθε δύο εβδομάδες, ενώ έπρεπε εγώ να παραδώσω το διαβατήριό μου και ενώ δεν μπορούσα να δουλέψω τις εβδομάδες που είχα το παιδί μαζί μου. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Ο, άντρας μου, ο πρώην άντρα μου όμως, και αφού απεδείχθη ότι απαράνομα είχε πάρει το παιδί, δεν είδε καμία συνέπεια. Εκτός από το τώρα που έχουμε πια φύγει, που δεν έχει το γιο του, ενώ εγώ έχω χάσει τα πάντα. Όταν είχε πάρει το παιδί μου, έχασα και τη δουλειά μου ακόμα, ε, την καριέρα μου, το παιδί μου. Ε, προσπάθησα να συνομιλήσω με τον πρώην άντρα μου, αλλά δεν δέχτηκε να διαπραγματευτεί μαζί μου και δεν καταλάβαινα ίσως μέχρι τώρα το συνέβαινε, γιατί ίσως να μην ήταν τόσο ε, ευφύης ο πρώην άντρα μου και δεν κατέφυγε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δανίας για να κάνει άλλη μία ψευδή καταγγελία εις βάρος αλλοδαπού, mm. Ναι. γιατί αν το είχε κάνει αυτό θα ήταν τελείως διαφορετικές εξελίξεις. Τώρα γύρισα στην πατρίδα μου, έχω αρχίσει να ξαναχτίζω το σπιτικό μου, δεν μπορώ να... Ε, πω ότι ε, παραπονιέμαι, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν μπορώ να ξεχάσω και τόσα πέρασα στη Δανία. Όπως ε, διαπιστώνει στα συμπεράσματα της υπόθεσής μου η Επιτροπή σας, συμπληρώνει ότι η Δανία είναι και συμβαλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ω εκ τούτου υποχρεούται να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, συγκεκριμένα δε και το δικαίωμα σε μια οικογενειακή ζωή. Η Δανία όμως δεν έκανε σεβαστά τα δικά μου, αλλά ούτε και το παιδί μου τα δικαιώματα όταν βρισκόμασταν στη Δανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαρή Κατλίν Τενής, Αρς Άσπελιν. Ευχαριστώ πολύ. Αναφορά η παριθμόν 28. Κυρία Οξάνα Τζούλ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω έρθει εδώ προσωπικό σήμερα για να κάνω μία δήλωση με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει να σταματήσουν οι παραβιώσεις των δικαιωμάτων των αλλοδαπών γυναικών και των παιδιών στη Δανία. Όπως συνέβη στη Βικτόρια και σε μένα. Με το που γεννήθηκε η Βικτόρια άλλαξε συμπεριφορά ο άντρα μου, πρώην άντρα μου ε, και άρχισε να με φέρεται βάναυσα. Μου απαγόρευε να επισκέφτομαι την οικογένειά μου στη Ρωσία ούτε καν δεν μπόρεσα να δείξω το παιδί στην ε, Ρωσίδα γιαγιά της, ενώ ήταν και εκείνος πιο κεκλημένος να έρθει μαζί. Μας, ε, ε μου έκρυψε τα, το, το πιστοποιητικό γεννήσεως της κόρης μου, δεν με άφησε ούτε καν αντίγραφό του να κρατήσω. Ε, κακοποιούσε το παιδί ταράζοντάς το, κρατώντας το από τα πόδια κρεμασμένο με το κεφάλι κάτω, λέγοντας ότι αυτός είναι ένας τρόπος να αναπτυχθεί η ευφυΐα του παιδιού. Απειλούσε ότι θα με απελάσει με τη βοήθεια του, ε, του, του Δήμου, του Δημοτικού Διαμερίσματος που μέναμε στη Δανία και στο τέλος άρχισε να με απειλεί ότι θα εξαφανιστεί μαζί με τη Βικτόρια και άρχισε να πετάει τα πράγματά μου έξω από την πόρτα λέγοντας μου ότι πρέπει να φύγω από το σπίτι. Ήταν 1,5 έτους η Βικτόρια όταν χρειάστηκε να καταφύγουμε σε ένα άσυλο για κακοποιημένες ε, γυναίκες και παιδιά. Όταν ήταν δύο ετών όμως η Βικτόρια το 2010 μου αφαίρεσαν την επιμέλειά τη με λόγο μόνο ότι προσπάθησα ε, με, με, με, μόνο επιχείρημα αυτά που προέβαλε ο πρώην, ο πρώην σύζυγός μου, ο δανός σύζυγός μου στο σύστημα της Δανίας. Με μόνο επιχείρημα δηλαδή ότι είμαι Ρωσίδα, ότι όλοι οι συγγενείς μου είναι στη Ρωσία και ότι φοβάται πώς θα πάρω τη, τη Βικτόρια στη Ρωσία. Από το 2010 και μέχρι σήμερα δεν έχω την επιμέλεια του παιδιού το οποίο βλέπω μόνο πέντε μέρες κάθε δεκαπενθήμερο, ενώ εκείνος το κρατάει τις υπόλοιπες εννέα μέρες. Η πρώτη απόφαση του Δανέζικου Δικαστηρίου αναφέρεται σε μία έκθεση εισήγηση ειδικού εμπειρογνώμονα για θέματα παιδιών, ο οποίος συνιστά το παιδί, ε, την επιμέλεια του παιδιού να πάρει αποκλειστικά ο πρώην σύζυγός μου, Δανός, με επιχείρημα ότι είναι συναισθηματικά πιο προσκολλημένο στο δανό πρώην σύζυγό μου το παιδί. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι η κόρη μου εκείνη την εποχή ήταν μόλις δύο ετών και ότι ακόμη τη, θύλαζα. Και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να είναι συναισθηματικά πιο προσκολλημένη στον πρώην σύζυγο. Και άλλα δικαστήρια στήριξαν τις αποφάσεις τους στα ψέματα του πρώην ε, συζύγου ότι τάχα δεν συνεργαζόμουν σε θέματα που αφορούν τη Βικτόρια και χωρίς άλλες αποδείξεις μόνο και μόνο επειδή είμαι άλλο δαπή. Εγώ επέδειξε καλό πνεύμα συνεργασία σε σχέση με τη Βικτόρια. Έχω έκθεση από το παιδικό σταθμό ότι ήμουν παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις σε όλα τα θέματα που αφορούσαν τη Βικτόρια ή τις επισκέψεις σε γιατρούς, ότι συμφωνούσαμε σε διάφορα πράγματα ε, σε σχέση με, το, με τη Βικτόρια, ακόμα και για την επιλογή του σχολείου που θα πήγαινε αργότερα. Δεν υπάρχει ουδεμία αίτηση στην Stats for Falting ή σε άλλες αρχές ε, κοινωνικής πρόνοιας που να ε, αποδεικνύουν πως δεν συνεργάστηκα εγώ σε θέματα που αφορούν την κόρη μου και, παρα, και εκτός του ότι με ουστέρισαν την επιμέλεια της χώρας μου και της χορίσμου μου και περιόρισαν και το δικαίωμα να την επισκέπτομαι και να τη βλέπω, οι αρχές της Δανίας, οι Stats for Valting, έχουν απαγορέψει και να πάω διακοπές στη Βικτόρια σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός Δανίας. Δεν μου επετράπει τον Ιανουάριο που θέλω να την πάρω διακοπές τώρα, το, το Δεκέμβριο αυτόν του 2013 ήθελα την πω αλλά δεν μου επιτράπει. Και αισθάνομαι ότι βρίσκομαι φυλακή εδώ στη Δανία. Δεν αξίζω αυτή την αντιμετώπιση. Είμαι μορφωμένη γυναίκα, αξιοπρεπής και έντιμη. Είμαι καλή μητέρα και έχω δικαίωμα και εγώ όπως και η κόρη μου σε μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ να επιτρέψετε να βοηθήσετε να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση στην επιμέλεια με την κόρη μου, με δικαίωμα σε επισκέψεις και με δικαίωμα να καπερνάμε τι εκοπές μας και έξω από τη Δανία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει κύριε Παλιαδέλη. «26 τώρα. Άννη Νίλσεν. Είσαστε εδώ κύριε Νίλσεν. Στη δική μου περίπτωση έχει υπάρξει παραβίαση της σύμβασης της Χάγης και των παιδικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ο ΙΕ. Πρόκειται για δύο παιδιά μικρής ηλικίας, κάτω των 8. δεν έχουν ενδιαφερθεί για τα συμφέροντα των παιδιών μου διότι δεν είναι εθνοτικός δανή. Και η αντιμετώπιση από τις δανέζικες αρχές δείχνει ότι υπάρχει συστηματική άνηση μεταχείριση. δεν εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Δανέζικη κυβέρνηση για την προστασία των ανθρωπίνων και παιδικών και γονικών δικαιωμάτων. Ε? Έχει παραβιαστεί επίσης και η σύμβαση που ισχύει στη Δανία για την ιδιωτική ζωή. Δεν με πληροφόρησαν, δεν μου δώσαν πρόσβαση σε όλους τους φακέλους που με αφορούσαν. μου συμπεριφέρθηκαν σαν να είχα κλέψει τα παιδιά μου, σαν να τα είχα απαγάγει. Ενώ τα άρθρα, το άρθρο 6 της Συνθήκης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έγινε σεβαστό και αυτά οφείλονται όλα στην τεράστια παραπληροφόρηση του πρώην άντρα μου. Ζήτησα λοιπόν διαμεσολάβηση πριν πάμε στο δικαστήριο. Αλλά στάλθηκε μία αίτηση στο Δανέζικο Δικαστήριο που δεν ήταν σωστά συμπληρωμένη και γι' αυτό τα δανέζικα δικαστήρια δεν έκαναν έρευνα όπως ήταν υποχρεωμένα πριν δώσουν τα παιδιά μετά από 14 μήνες στον πατέρα τους. Όλα τα έγγραφα που στάλθηκαν από τον Υπιαγωγείο, από τους ψυχολόγους, από το Δημαρχείο δεν ελήφθησαν υπόψη. Τα δικαιώματα των παιδιών μου λοιπόν να ζουν ε, με τη μητέρα τους έχουν παραβιαστεί. Εκτός αυτού δεν έλαβα ποτέ επιστολή από το δικαστήριο τον Αύγουστο του 11 που να μου λέει ότι ε, που να με πληροφορεί. Και εγώ σοκαρίστηκα και τα παιδιά μου. Είχα μόνο δύο μέρες για να προετοιμάσω τα παιδιά μου για επιστροφή στην Ιταλία χωρίς τη μητέρα τους. Διότι η εγγύηση που υποσχέθηκε ότι θα έκανε ο πρώην σύζυγός μου να μην συνεχίσει δεν είναι δεκτή, δεν, δεν στάλει ποτέ. Εκτός αυτού το δικαστήριο αρνήθηκε μετά από έξι μήνες όταν θα επέστρεφα στην Ιταλία να δεχτεί να δω τα παιδιά μου. Επίσης παραβιάστηκε η συνθήκη της Χάγης στο άρθρο 13β. Τα παιδιά έμειναν στη Δανία πάνω από 14 μήνες. Ο πατέρας τους μιλούσε μόνο Ιταλικά και εκείνα μόνο Δανέζικα. Τα παιδιά ήταν τότε τριών και πέντε ετών και ε, τα φρόντιζαν γυναίκες άσχετες από μένα και από τον πατέρα τους. Έτσι τραυματίστηκαν ψυχολογικά και αυτά τα έχουν καταγράψει επαγγελματίες. Προσπάθησα να πάρω απαντήσεις και βοήθεια από τις δανέζικες αρχές, αλλά ό,τι και να έκανα έπαιρνα αρνητική απάντηση. Ζήτησα επίσκεψη και μου απαντούν δεν βλέπουμε κανένα λόγο να συναντήσετε τα παιδιά σας ή να, με, να σας συναντήσουμε. Επίσης δύο φορές Ζήτησα στο, από το Δανέζικο Οικογενειακό Συμβούλιο να αναλάβει την υπόθεση, δεν το έκανε. Την τελευταία φορά απάντησαν το Σεπτέμβριο του 2013 ότι είχαν αποφασίσει να μην ερευνήσουν την υπόθεση, διότι έχει το δικαίωμα ως Δανέζος διαμεσολαβητής. Επίσης, έστειλα γράμμα σε Ιταλό δικηγόρο ζητώντας από τις Ιταλικές αρχές, από Ιταλό δικηγόρο, από τις και Αρχές να με βοηθήσουν οικονομικά γιατί είχα παγιδευτεί στην Ιταλία. Αλλά τελικά έχασα την κυδαιμονία των παιδιών μου και τελικά ο πρώην σύζυγός μου κατάφερε να πάρει τα παιδιά από μένα για πάντα. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή σας να βοηθήσετε και μένα και τα παιδιά μου ώστε να δοθεί η βοήθεια στην οποία έχουμε δικαίωμα ως δανείοι πολίτες, όπως οι δανείοι πολίτες. Επίσης ζητώ να ερευνήσετε αυτήν τη συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων γυναικών και παιδών. Ευχαριστώ. Now we move to... Πάμε τώρα στο 27. going to a statement from, Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω εγώ την παρουσίαση εκ μέρους κυρίας Χόρτης Άντελα Τόρτυρ, που δεν μπορεί να έρθει διότι φυλακίστηκε χθε μόλις. Ζουν σε φόβο και εκείνη και η κόρη της τα τελευταία χρόνια με τις ε, ε, με την κακοποίηση του πρώην συζύγου και πατέρα του παιδιού. Έφυγαν από το σπίτι, το Υπουργείο όμως τους είπε ότι αν θέλουν να επιστρέψουν στην Ισλανδία για να αποφύγουν αυτή την κακοποίηση ε, θα τους προσφέρει προστασία. Αλλά δεν συνέβη αυτό. Φυλακίστηκαν, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν εχθές στη Δανία χωρίς καμία ενημέρωση. Δεν έχει κανένα τρόπο να προσφύγει για να ζητήσει την προστασία της. Για πολλά χρόνια έχει ζήσει η ίδια και οι της σε καθεστώς τρόμο και ζητούν την υποστήριξή σας. Τη χρειάζονται πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα μας κάνετε την παρουσίαση της δικής σας αναφοράς της υπαριθμών 35. Αξιότιμα μέλη τη Επιτροπής, σας ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να μιλήσω σήμερα. Ο γιος μου ήταν πέρσι τον Απρίλιο τεσσάρων ετών. Γύρισε σπίτι και είδα σημάδια κακοποίησης από την πλευρά του πατέρα του. Κάναμε ό,τι προβλέπει ο νόμος, όπως μας είπαν άλλωστε στην Δανία, γιατί ζήτησα ενημέρωση ότι πρέπει να κάνω στο νοσοκομείο. Αλλά αρνήθηκαν οι αρχές να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση, ακόμα και η αστυνομία. Ε, δεν του μίλησαν ε, όμως του άντρα μου, δεν έκαναν τίποτα γιατί ήταν τεσσάρων ετών το παιδί μόλις και θεωρήθηκε ίσως όχι αξιόπιστος μάρτυρας. Πάντως εγώ χρειάστηκα, αναζήτησα περισσότερες πληροφορίες και πήγα σε ειδικό για τα παιδιά και ζήτησα να κοιτάξει το παιδί μου ε, ο ψυχολόγος να, για να πιστεί εάν λέει την αλήθεια. Λοιπόν, το ναι. παιδί μου πήγε πολλές φορές και την επισκέφθηκε και εκείνη πίστηκε ότι της λέει την αλήθεια. Σε μια έκθεσή της μας ε, βεβαιώνει ότι διαπιστώνει πως όντως πρέπει να έχει λάβει χώρα αυτή η κακοποίηση και ότι το παιδί μου πρέπει να προστατευτεί να μην επισκέπτεται τον πατέρα του. Ο πατέρας του όμως διεκδίκησε τα δικαιώματα αυτά επικοινωνίας με το παιδί και μας πήγε σε δικαστήριο επιβολής ε, των αποφάσεων ε, για να με αναγκάσει να του παραδώσω το παιδί. Πράγμα το οποίο εγώ δεν ήθελα να κάνω γιατί το παιδί μου υπέφερε πολύ και ήξερα ότι λέει την αλήθεια. Ωστόσο, οι αρμόδιε αρχέ δεν θέλησαν να του αφαιρέσουν το δικαίωμα επικοινωνία με το παιδί, διότι αυτό ισχυρίστηκε σε μια συνάντηση ότι ποτέ δεν έχει ακουμπήσει το παιδί και έτσι πίστεψαν τον πατέρα και όχι το παιδί που ήταν 4 ετών. Όταν έφτασε και η έκθεση του ψυχολόγου, ζήτησα από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν με προσοχή το τι έχει συμβεί. Και έτσι ζήτησαν από άλλον ψυχίατρο να παρακολουθήσει την ζωή μας για δύο μήνες για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Και το Δεκέμβριο καταλήγει η ψυχίατρος αυτή στο συμπέρασμα ότι η, επίσης, η επικοινωνία με τον πατέρα πρέπει να γίνεται μόνο για δύο ώρες και με επιτήρηση. Αυτό συνέβαινε από το Δεκέμβριο μέχρι τώρα και εντωμεταξύ αργόρασα πολύ ε, πλήρωσα ένα πολύ ακριβό τίμημα γιατί θέλησα να προστατέψω το παιδί μου. Βρέθηκα στη φυλακή για δύο μέρες, για έξι μέρες. Ε, μετά μόνο από έξι μέρες με αποφυλάκησε το δικαστήριο. Ελπίζαμε ότι στα τέλη Ιανουαρίου πια θα μπορούσαμε να ζήσουμε σε συνθήκες ειρήνης και ηρεμίας αφού είχε, δοθεί απόφαση, είχε εκδοθεί απόφαση για την επιτηρούμενη επίσκεψη, αλλά αμέσως μετά ξεκίνησε μια νέα διαδικασία για αποκλειστική επιμέλεια από πλευρά του πρώην συζύγου και γι' αυτό διερωτώ με γιατί εμείς πρέπει να ζούμε σαν πρόσφυγες, όπως οι Εβραίοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να κρυβόμαστε και αν θα πρέπει να περάσουμε από την ίδια ταλαιπωρία και πάλι αν υπάρχει κανείς που μπορεί να μας προστατέψει. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you as well. Και εγώ ευχαριστώ. Σημείο 38. Η κυρία Μη που προσπαθεί να διαφυλάξει την ε, να προστατεύσει την ταυτότητά της, να κρατήσει την κρυφή ταυτότητά της, ε, μας έχει στείλει ένα βίντεο για το οποίο δεν υπάρχει ήχος προς το παρόν, δεν ακούγεται τίποτα. problem, should I read it? Should I read her statement? I have a, I have a statement.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 Thank you very much for listening. No, this is too much, I think. Νομίζω ότι είναι μια μέρα που, μας, ε, που έχουμε μάθει για πράγματα πολύ συγκλονιστικά σήμερα. Θα δω μάλλον ένα βίντεο για το σημείο 40. Also wishing to preserve her ε, privacy.